Ζαλέσκη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Πολωνική Προεδρία θεωρεί ότι αυτή η, αυτό το νομοθέτημα για την προστασία στα ποινικά είναι εντάξει, ε, είναι κάτι το άρτιο, αυτό πρόκειται να σύντομα το γίνει το κοινοβούλιο σας. Τώρα, όσον αφορά την Προεδρία, έχουμε προσπαθήσει να προλιάνουμε το έδαφος και επίσης ε, είμαι θα ότι και η ε, δανεί συνάδελφοι θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση βεβαίως. Θεωρούμε ότι είναι θετικό το σχέδιο κειμένο, ευχαριστούμε γι' αυτό. Τώρα, στρέφουμε στους συναδέλφους. Κύριε Κέρχο, παίρνει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, πρώτα-πρώτα ξεκινώ αναφέροντά σα ότι βεβαίως και θεωρώ ότι πάρα πολύ θετική αυτή η πρωτοβουλία Ξέρετε ότι και στη χώρα μας διαλέξαμε να μην αυτοεξαιρεθούμε από τη σχετική νομοθεσία τον Αύγουστο δε τρέχοντος έτους και εμείς έχουμε να σας πούμε ότι μας ενδιαφέρει και δεν θέλω να μην παρεξηγηθεί σε γήτρια, διότι και εγώ είμαι νομικός εκτός από νομοθέτης. Έχω να της πω κάποια πια θέματα, ελπίζω λοιπόν να μην ε, παρεξηγηθεί, διότι με προβληματίζουν κάποια σημεία και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το οποίο τώρα μας απασχολεί, διότι θεωρώ ότι είναι προς το συμφέρον των θυμάτων, αλλά επίσης ε, αυτό είναι και προς το συμφέρον εκείνων οι οποίοι φύστανται την ε, ποινική δίωξη ως ε, ένοχοι, ως φερόμενοι ως ε, ένοχοι. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει μας τη λειτουργία της δικαιοσύνης και αυτό είναι πάντοτε η βασική μας η, η μέρη με τώρα. Όπως θα θυμάστε, όσον αφορά την νομοθεσία για προστασία στην ΕΟΚ, έχουμε ένα σωρό θέματα ποινικά, μια ολοκληρωτικά κατάλογο, αλλά και άλλα μη ποινικά που δεν είναι αναγκαστικά ποινικά δικήματα ή στα κράτη-μέλη. Αυτά στην οδηγία για την εντολή προστασίας. Και τα θέματα προστασία προστασίας σε κάποιες χώρες καλύπτονται από τα πολιτικά δικαστήρια. Βλέπετε επομένω τι, τι εγχείρημα έχουμε μπροστά μα. Οπότε, τι γίνεται σε περίπτωση ανθρωποκτονία, είναι ποινικό ή αστικό. Εδώ έχουμε και το θέμα ε, της, ε, του, του διπλού ποινικού χαρακτηρισμού. Και αν κάποιος λοιπόν ποινική δίωξη για κάποιο αδίκημα, ε, εμπλέκεται και στις δύο διαδικασίες, και στην πολιτική και στην ποινική. Και, εδώ υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει διαφορετική αντιμετώπιση σε κάθε διαδικασία, στην πολιτική και στην ποινική. Θα, θα να είναι αυτονόητο να νομίζω ότι οποτεδήποτε κανείς τα ανακατεύει τα πράγματα Α, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο background για τέτοιες συζητήσεις η μουσικούλα. Όποτε επομένως προκύπτει. Α, να βλέπω πω, και, και καμπάνες, ηχούν καμπάνες. Κυρία Πρόεδρε, σας παρακαλώ κάντε κάτι, να έχουμε μουσικούλα, να μας συνοδεύει στις συζητήσεις μας Ιού. Ναι, ναι, ναι, στα, στα κτηνοτροφία. Παίζουν στι αγελάδε ε, μουσικούλα για να παράγουν περισσότερο γάλα. Λοιπόν, τι έλεγα. Ότι οποτεδήποτε προκύπτει τέτοιο ανακάτεμα, μπορεί να το βεβαιώσει οποιοδήποτε νομικό συμβεί στην αίθουσα. Θα καταλάβαινε τι εννοώ που λέω για το ανακάτεμα. Το να ανακατεύουμε τα αστικά θέματα με τα ποινικά, αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε ατυχή αποτελέσματα. Να, Φερρυπίν, θυμάμαι κάποια θέματα που έχουν σχέση και με το φορολογικό δίκαιο. Πρέπει επομένω να δούμε πώς θα ξεκαθαρίσουμε τους χαρακτηρισμούς. Ας πούμε, σε κάποιες χώρες το να παρακολουθεί κάποιον ε, είναι ποινικό δίκημα. Το να ακολουθεί κάποιον ε, είναι δίκημα. Όλα αυτά όμως πρέπει να διευκρινιστούν περισσότερο. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουν. Τέλο πάντων, εγώ βλέπω πάρα πολύ θετική αυτή την προσπάθεια και η κυβέρνηση τη χώρα μου επίση ε, για να διαλέξει να συμμετάσχει τη αρέσει. Οπότε, ναι, ναι, στο κείμενο. Όμω, παρακαλώ, θα θέλω ασφαλώς τώρα στην επόμενη φάση που θα διεκπαιριώσουμε αυτό το κείμενο θέλω να κάνετε αυτά τα οποία σας είπα, να ξεκαθαρίσουμε περισσότερο αυτά τα ζητήματα. Το τι γίνεται, πού αρχίζει και πού τελειώνει η ποινική διαδικασία, πού αρχίζει και πού τελειώνει η πολιτική διαδικασία και κατά πόσον υπάρχει ένα μπέρδεμα, κατά πόσον υπάρχει κάποιο είδου επιρροή τη μια δικαδία στην άλλη και να εξασφαλίσουμε το ότι δεν θα παραβλάβουν τα δικαιώματα κάποιου ο οποίο ενδεχομένω υφίσταται ποινική δίωξη ε, γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αλλιώ νομίζω ότι δικαίω θα ενίστανται οι δικηγόροι για τα δικαιώματα του πελάτου τους. Οπότε θα μπερδευτεί πάρα πολύ το πράγμα αρκετά, ιδίω σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες. Αλλά πέραν όλων αυτών, ε, κυρία Πρόεδρε, γενικά το βλέπω θετικά. Όμως θα πρέπει το θέμα το εξετάσουμε με περισσότερη προσοχή. Ευχαριστούμε κύριε Κέρκοπ. Ο κύριος Φως. Ευχαριστώ. Εγώ γενικά υποστηρίζω αυτό το θέμα. Εσύ δηλαδή είναι η σωστή. Αλλά και εγώ έχω παρόμοιες ε, ανησυχίες όπως οι σκέψεις που εξέφρασε ο Τίμωθη Κέρκοπ. Δηλαδή εδώ προσπαθούμε να παραμείνουμε σε μια συστηματική δικαίου, ένα διαχωρισμό μεταξύ ε, ποινικού και αστικού δικαίου. Μήπως γίνονται ε, κάποια βήματα προς τα πίσω σε σχέση με την αναγνώριση στα επιμέρους κράτη. Η αναγνώριση, κατά τη γνώμη σας, είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολύ πολύπλοκο. Δηλαδή, όταν προτείνουμε κάτι χρειάζεται μετάφραση, χρειάζεται, χρειάζονται πολλά βήματα και ίσως ενδεχομένως υπάρχει κάποια άλλη λύση ώστε τα μέτρα προστασίας να είναι απλούστερα, να μπορεί το θύμα να αναγνωρίζεται πιο εύκολα. Όταν έχουμε ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, να έχουμε δηλαδή ένα απλούστερο και πιο άμεσο μέτρο. υπάρχουν ε, διαφορές όταν το δικαστήριο στη μία χώρα καθορίζει ε, κάτι το οποίο στην άλλη χώρα δεν υφίσταται ως μέτρο αυτό καθεαυτό. Εγώ θα ήθελα να ξέρω τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να είναι πιο άμεση η αναγνώριση. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Γκρίσμπαχ. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Θέλω και εγώ να συγχαρώ τον εισηγητή ε, για το έργο του, ε, την εισηγήτρια για το έργο της, που είναι πολύ, ε, φαίνεται ότι είναι πολύ απλή αυτή η έκθεση, αλλά είναι πολύ πολύπλοκη όσον αφορά την αποτελεσματικότητά της επιτόπου. Θα έπρεπε ήδη από το πρώτο κείμενο της οδηγίας να υπάρχει η αναγνώριση και ε, ελπίζω σήμερα να μπορέσουμε να οργανώσουμε την προστασία των θυμάτων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Επικράτεια. Ίσως να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες εφαρμογής, αλλά ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να τις ξεπεράσουμε. Ε, θέλω να υπενθυμίσω ότι περίπου 75 εκατομμύρια Ευρωπαίοι υφίστανται ε, τέτοιες παραβιάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και θέλουμε να παράσχουμε προστασία σε αυτά τα θύματα. Το κείμενο το έλαβα σήμερα το πρωί μόνο και δεν έχω προλάβει να το δω εις βάθος, άρα θα ήθελα μέχρι τις 29 Νοεμβρίου να το δω καλύτερα και επιφυλάσσομαι για τις τροπολογίες που ενδεχομένως θα υποβάλλω. Ε, σχετικά με την ταχύτητα της ε, προστασίας ε, υπάρχει ένα ζήτημα. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα νέο μοντέλο για τα πιστοποιητικά προστασίας που εκδίδονται, ούτως ώστε οι διαδικασίες ε, να διευκολύνονται στα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες λεπτομέρειες που ίσως πρέπει να διευκρινίσουμε γιατί το θέμα είναι εξορισμού πολύπλοκο. Μέχρι τις 29 του μηνός ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να επεξεργαστούμε περισσότερο αυτό το θέμα και χαίρομαι και για αυτά που άκουσα από την εισηγήτρια αλλά και από την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το ότι επιζητούν συνέπεια μεταξύ των κειμένων ούτως ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες εγγύησει και ο συντονισμός μεταξύ τη οδηγία και του κανονισμού. Τέλο πάντων, μέχρι τι 29 του μηνό, η ομάδα μου θα έχει τη δυνατότητα ε, να επιφέρει περαιτέρω διευκρινήσεις μέσω των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και στρέφομαι και πάλι στην εισηγήτρια, αν δεν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι. Κυρία Ρομέρο Λόπε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ εξετίμησα τα όσα είπε το Συμβούλιο αλλά και η Επιτροπή και κατά δεύτερο λόγο τώρα ξεκινούμε αυτή την ε, διαδρομή για την οποία επίσης θα ο κύριος Κέρκοπ είναι πάνω και στο η κυρία ε, Γρίσπερ και ο κύριος Φως μια που το θέμα εδώ είναι δύσκολο, οπότε όσο περισσότερη βοήθεια έχουμε για το κείμενο, τόσο καλύτερα θα τα καταφέρουμε για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο θέλουμε. Όντως, ο κ. Κέρχοπ έχει δίκιο που μας είπε για αυτή την αλληλεπίδραση η οποία ε, υπάρχει, διότι ακριβώς είναι το θέμα το οποίο συζητήσαμε για την ε, οδηγία που αφορούσε την προστασία. Όντω. αλλού υπάρχουν θέματα ποινικού δικαίου, αλλού τα ίδια θέματα εμπίπτουν στο αστικό δίκαιο. Θα πρέπει όμως τώρα να επεξεργαστούμε το ότι παρά το ότι έχουμε επομένω περιπτώσει που να συντρέχει το, το, το, το, αστικό δίκαιο, να πρέπει ταυτόχρονα με κάποιες τροπολογίες να φροντίσουμε για τα θέματα που εμπίπτουν στο ποινικό δίκαιο. Και είμαι σίγουρος ότι ο κύριος ε, Κέρκο πρόκειται να προετοιμάσει κάποιες τέτοιε τροπολογίες και το κείμενο θα βελτιωθεί. Ε, Βεβαίω και το θέμα είναι το τι προσέγγιση θα γίνει στην ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό. Βεβαίω και έτσι έχουμε την πιο διεκπαιρεωτική, πιο γρήγορη διαδικασία και για αυτό το λόγο θα λάβω υπόψη και αυτό το οποίο ο κύριος Φως σε σχέση με αυτό το, το, το, το, το νομοθέτημα, να το, πώς θα το βελτιώσουμε αυτές τις τροπολογίες. Είπε και η κυρία για να δούμε πώς αυτό το θέμα θα αντιμετωπιστεί καλύτερα, διότι το αξίζει. Και μας είπε ότι μας είπε ο κύριο Κέρχοπ σε σχέση με το όταν έχει προβλήματα διανοητικά, διανοητικά είπε ο ένοχος ας πούμε. Πώς θα ληφθούν κάποια μέτρα ασφαλιστικά, κατασταλτικά. Όμως αυτό θα προκύψει εκ των υστέρων αν έχετε προβλήματα διανοητικά, αυτός ο οποίος ε, επιτίθεται, αυτός ο οποίος ε, είναι ο θήτης, ας πούμε, θα πρέπει να κρατηθεί μακριά από το θύμα, αν επομένω είναι διανοητικά ασθενής. Αυτό θα πρέπει να συμπληρώσουμε και να ε, δούμε πώς μπορούμε να το ρυθμίσουμε με κάποια τροπολογία, γιατί τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο βεβαίως και επιδέχεται βελτίωση στο κείμενο, έτσι, με αυτά που είπαμε. Τώρα, έχουμε δεδομένο το κείμενο της Νομικής Επιτροπής σε σχέση με κάποιους ανηλίκους. Πάντως, εδώ είναι θέμα το οποίο μπορούμε να το προχωρήσουμε, έχουμε τα χρονικά περιθώρια και έτσι να είναι όσο γίνεται αρτιότερο το κείμενο. Σας ευχαριστώ. Ρομέρο Λόπες. Κυρία μου, θα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι 29 Δεκάτου εκπνέει η προθεσμία η σχετική με τις τροπολογίες. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα. Τι άλλο λέει η μερσία μας διάταξη. Όροι και προϋποθέσεις ισόδια δημονισμικών τριτών χρόνων στο πλαίσιο της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης. Σαλβατόρα Ιακολίνο είναι ο συγγητής. Και έχει διανύμει κάποια κείμενα συμβιβαστικών τροπολογιών. Νομίζω τα έχετε πάει. Θα δώσουμε πρώτα πρώτα τον λόγο στον κύριο Γιακολίνο για αυτές τις τροπολογίες και στη συνέχεια να μας πει και το Συμβούλιο πώς έχουν γίνει τα πράγματα δώσουν το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίω και στου συναδέλφου, όποιον θέλω Κύριε Γιακολίνο, είδε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όσον αφορά το ζήτημα αυτό που έχουμε στη μερίσια διάταξη, ξέρετε ότι ε, κάναμε πολλές συνεδριάσεις και στα πλαίσια της Επιτροπής μας, αλλά και αλλού. Μιλήσαμε με τους σκιώδεις ηγητές των πολιτικών ομάδων και στην τελευταία μας συνεδρίαση που έγινε πριν από μερικές μέρες συνεδριάσαμε για το ζήτημα αυτό, στο Στρασβούργο συγκεκριμένα. Σε ορισμένε περιπτώσει οι σκιώδει συγητές δεν ήταν σε θέση να έρθουν στι συνεδριάσει Πάντως ε, είχα τη δυνατότητα να συνομιλήσω με τον συνάδελφό μου, ο οποίο συντάσσει τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης. Έχουμε καταλήξει λοιπόν σε 21 συμβαστικές τροπολογίες, οι οποίες εστάλησαν στους συναδέλφους και τους κάλεσα βέβαια να κάνουν στη συνέχεια παρατηρήσεις και σχόλια. Και προσπαθήσαμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο μέτωπο, στο μέτρο του δυνατού. Είμαι επίση σε επαφή βέβαια με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Οι συμβαστικέ τώρα τροπολογίε αντικατοπτρίζουν κάποιε από τι σκέψει τι οποίε εκφράσαμε κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεών μας, ιδίω για του ορισμού για το άρθρο 50 για παράδειγμα, το οποίο απαιτεί από εμά να καθορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μία πιο ενιαία προσέγγιση μαζί με την Επιτροπή Απασχόλησης είναι άλλωστε και το σημείο αυτό του κειμένου, το οποίο άπτεται και των δικών τους αρμοδιοτήτων, εφόσον πρέπει κανείς να καθορίσει τους εργοδότες, τους εργαζόμενους, τους εμπειρογνώμονες. Έχουμε καταφέρει λοιπόν να καταλήξουμε σε συμφωνία όσον αφορά την χρήση των ορισμών, όσον αφορά για παράδειγμα τον ορισμό για την μπλε κάρτα όσον αφορά τους εμπειρογνώμονες, τους ειδήμονες και στην ίδια προσέγγιση έχουν προχωρήσει και για το ζήτημα της ενίας άδεια. Προσπαθήσαμε επίσης να συμφωνήσουμε και για την απέτηση να προβλέπεται πρόσβαση και δυνατότητα κινητικότητας μεταξύ κρατών εκτός και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στις χώρες αυτές. Επίσης, ε, όσον αφορά τις συλλογικέ συμβάσεις, ασχοληθήκαμε και με αυτές. Προβλέπεται μία περίοδος 9 μηνών για τους managers, τριών μηνών για τους ασκούμενους. Έχουμε επίσης προβλέψει ένα νέο χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις κυρώσεις κάθε φορά που μπορεί να παρουσιάζονται προβλήματα με τους εργαζόμενους. Θέλουμε επίσης να διευθετήσουμε ζητήματα οικογενειακής φύσης. Κάθε φορά που ένας εργαζόμενος πρέπει να αλλάξει τόπο εργασίας. Και επίσης είπαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και ένα κοινό χρονοδιάγραμμα, μια κοινή χρονική περίοδος όσον αφορά το ζήτημα της άδειας παραμονής. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα όσον αφορά το ζήτημα της υγειονομικής ε, κάλυψης του της συζύγου του εργαζόμενου. Πρέπει λοιπόν να προβλέπετε μια τέτοια παροχή, μια τέτοια κάλυψη από τα κράτη-μέλη. Υπάρχει βέβαια και ένα σημαντικό ζήτημα επικουρικότητας ως προς αυτό. Όσον αφορά την κινητικότητα μεταξύ των κρατών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, προβλέπεται ήδη ένα σύστημα γι' αυτό. Είχαμε πολλές παρεμβάσεις και είπαμε ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζομένων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες, προασπίζοντας όμως και τα συμφέροντα των ήδη φυσταμένων εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχουμε διακρίσεις μεταξύ των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να ισχύει ένα καθεστώ ούτε διακρίσεων ούτε προνομίων. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση στην εργασία, ισότιμε αποδοχέ αποδοχές και να μην υπάρχει βέβαια καμία περίπτωση διάκριση μεταξύ εργαζομένων χώρας προέλευσης και χώρας υποδοχής. Η εργασία που είχε γίνει μέχρι στιγμή ήταν ιδιαίτερα θετική, ιδιαίτερα ενθαρρυντική δεν έχουμε καταφέρει βέβαια να διευθετήσουμε όλα τα κρεμή ζητήματα. Ελπίζουμε πάντως ότι πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να εργαστούμε βάσει των 21 αυτών συμβαστικών τροπολογιών και να καταλήξουμε τελικά σε ένα κείμενο το οποίο θα χαίρει αν όχι ομοφωνία, τουλάχιστον μιας ευρύτατης υποστήριξης. θέλουμε μέσω του κειμένου αυτού να επιτρέψουμε και στους ε, εργαζομένους που έρχονται από τρίτες χώρες να υποφεληθούν των ε, εργασιακών συνθήκων πισχύνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά αυτόν τον τρόπο όμως να υποφεληθούν και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να έχουμε μια σημαντικότερη οικονομική ανάπτυξη μέσω των νομοθετημάτων αυτών, ιδίω την δύσκολη αυτή, δυσχερή οικονομικά περίοδο που διανύουν οι επιχειρήσει και οι ευρωπαϊκέ οικονομίε. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή μα, τη Γραμματεία τη Επιτροπή μα, όλου του συναδέλφου με του οποίου συνεργάστηκα. Να ευχαριστήσω επίση και το Συμβούλιο, καθώ επίση και τι Προεδρίε Συμβουλίου, παρελθούσε και φυστάμενε. Ολοκληρώνω στο σημείο αυτό, κυρία Πρόεδρε, και είμαι στη διάθεσή σας για να ακούσω και τις παρατηρήσεις των συναδέλφων και ελπίζω ότι οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες ουσιαστικά θα διευκολύνουν την εργασία μας και ελπίζω θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε σύντομα. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Το λόγο τώρα έχει η Πολωνική Προεδρία, κυρία Σκύμπα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μέχρι τώρα έχουν γίνει τρεις συνεδριάσεις της σχετικής ομάδος εργασίας στο Συμβούλιο και ασχολούμεθα με τη σχετική οδηγία. Και μάλιστα σήμερα, την ώρα που μιλάμε, γίνεται μία σχετική συνεδρίαση και την επόμενη εβδομάδα θα γίνει άλλη μία συνεδρίαση για την ίδια οδηγία. Και επειδή ορισμένα θέματα πρέπει να συζητηθούν σε υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, το περασμένο μήνα συζητήθηκαν δύο θέματα στη συνεδρίαση της Επιτροπής Στρατηγικής για το Άσυλο. Συζητήθηκε το πεδίο εφαρμογή της οδηγίας, καθώς και η βραχυπρόθεσμη κινητικότητα. Την επόμενη εβδομάδα στις 30 η ίδια Επιτροπή θα ασχοληθεί με τους ορισμούς τους ορισμούς που ανέφερε και ο εισηγητής. Τώρα όσον αφορά την κατάσταση στο Συμβούλιο και τα τρία βασικά θέματα, χρειάζονται ακόμη κάποιες εξηγήσεις. Το πρώτο ζήτημα είναι οι ορισμοί. Πρέπει να αποφασίσουμε αν θα επιλέξουμε τους ορισμούς όπως έχουν οριστεί από το GATS, ή αν θα παραμείνουμε στους ορισμούς που έχουμε τώρα στο κείμενο, γιατί τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις επί του θέματος. Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ορισμένα κράτη-μέλη πρόσφατα υπέβαλαν μία πρόταση για τα άτομα που ουσιαστικά μένουν έξω από την οδηγία. Δεν πληρούν τις διατάξεις εισόδου ως υπάλληλοι στον τομέα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Και αυτά τα κράτη-μέλη ζητούν κάποια διαφορετική λύση που να τους παρέχει κάποιο περιθώριο ελιγμών. Δηλαδή να βρεθεί μια λύση για τα άτομα αυτά που δεν προέρχονται από τον τομέα της πληροφορικής και των επικοινωνιών. Θα είναι σχεδόν παρόμοιο το καθεστώς τους. Και το Συμβούλιο υποστηρίζει μια τέτοια λύση του να είναι σχεδόν παρόμοιο με αυτά τα άτομα. Ένα άλλο θέμα αφορά την κινητικότητα περιορισμένου χρονικού διαστήματος. Εδώ υπάρχει ειδική πλειοψηφία για την κινητικότητα μέχρι τρεις μήνες, όπου προτείνεται να προσφέρονται η μεγαλύτερη δυνατή πρόσβαση στους εργαζόμενους στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για να μην επιβαρύνονται με περιττές διοικητικέ επιβαρύνσεις. Περιμένουμε τις επόμενες δύο συνεδριάσεις ε, με περισσότερες διευκρινήσεις και θα γίνουν ε, και άλλες συναντήσεις με τους εισηγητές για να μπορέσουμε το συντομότερο δυνατόν να σας ενημερώσουμε για την πρόοδο στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ και στρέφομαι στην Επιτροπή, κυρία Σμιτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Γιακολίνο, για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε και τώρα όπως και στο παρελθόν. Ελπίζω ότι θα καταστεί δυνατόν ε, να συμφωνήσουμε για μια οδηγία φιλόδοξη, η οποία ε, προσπαθεί να καταλήξει σε εναρμόνιση για τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις. Προς το παρόν ε, δεν μπορώ να σας δώσω τις αντιδράσεις μας για τις τροπολογίες. Ε, λίγο πολύ συμβαδίζουμε το στόχο της οδηγίας, δηλαδή θέλουμε να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και να βελτιώσουμε την κατάσταση όσον αφορά την τεχνολογία πληροφορική και επικοινωνιών. Για τους ορισμούς, όπως έχουμε ήδη πει, θέλουμε να έχουμε ορισμούς αρκετά ευέλικτου, που όμω να μην είναι αμφίσιμοι. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν είναι υψηλή ειδίκευση και κάτοχοι μπλε κάρτα οι εργαζόμενοι στον τομέα αυτό. Αυτό το έχουμε κατά νου. και για την επανένωση των οικογενειών ίσως είναι πολύ περισσότερο ε, φιλόδοξο αυτό που προτείνεται και για την ίση μεταχείριση η Επιτροπή ε, έχει προτείνει να ισχύουν οι κανόνες που ισχύουν και για τους αποσπασμένους εργαζόμενους. Αυτοί να ισχύουν και για τους εργαζόμενους στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών που μετατίθενται ενδοεπιχειρησιακά. Επαναλαμβάνω ότι η Επιτροπή επιθυμεί μια φιλόδοξη οδηγία και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή της. Δηλαδή όσοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας μπορούν να την χάνουν διαφορετικών αδειών που δεν θα είναι άδειε ε, ICT αλλά αν κάποιος δεν πληρεί τα κριτήρια που προβλέπονται στην οδηγία θα πρέπει να δούμε αν θα εμπίπτει σε ένα εθνικό σύστημα και όχι να καλύπτεται από την οδηγία. Αυτό θα δημιουργούσε παράλληλα συστήματα και θα ήταν κατά της εναρμόνισης. Η κινητικότητα εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα σημαντικό θέμα και αποτελεί και προστιθέμενη αξία της παρούσα οδηγίας. Αν αποδυναμώσουμε την κινητικότητα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν πληρείται ένας από τους στόχους της οδηγίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σμιτ. Ας ξεκινήσουμε τη συζήτηση τώρα και θα δώσω το λόγο στην κυρία Γιακονσάρη, που είναι η συγγήτρια στην Επιτροπή Απασχόλησης. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τους εξαιρετικούς διερμηνείς μας, οπότε μου μιλήσω στα φιλανδικά. Λέω μιλήτρια. Έχω να σας πω ότι πρόκειται για κάποιο περίπλοκο θέμα, πρόκειται για δύσκολο νομοθέτημα. Και εδώ πέρα έχουμε από κοινού δεσμευτεί και η Επιτροπή των Ελευθεριών αλλά και η, πολιτική, και η Επιτροπή της Απασχόλησης ούτως ώστε να ρυθμιστεί αυτό το θέμα διότι συνολικά πρόκειται για μια πάρα πολύ θετική προσπάθεια πρόκειται για κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με τη στρατηγική την Ευρωπαϊκή Ενόψη του 2020 και ότι θέλουμε επομένως να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους ε, κατηρτισμένους από τρίτες χώρες και θα πρέπει να δούμε πώς δεν θα μας υπονομεύει η γραφειοκρατία. Όμως θα πρέπει να λύσουμε και κάποια βασικά προβλήματα και κατά τη γνώμη μου εδώ ένα βασικό πρόβλημα πρόβλημα είναι ότι έχουμε τώρα ένα σωρό διαφορετικούς ε, τρόπους ούτως ώστε να βοηθήσουμε την κινητικότητα και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τους ανθρώπινους σπόρους. ε, πώς θα μπορέσουμε να δούμε ε, τι θα γίνει με την οδηγία ICT και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σαν μια δέσμη μέτρο, σαν ένα σύνολο, σαν ένα πακέτο. Τώρα, Όσον αφορά τώρα του ορισμούς η Επιτροπή Απασχόληση επίση εξετάζει το θέμα, να δούμε πώς θα βρεθεί ένας συμβασμό, γιατί είναι πάρα πολύ βασικό οι ορισμοί να μην είναι πάρα πολύ γενικόλογοι και δεν θα πρέπει να ανοίξουμε ένα παράθυρο, ένα χάσμα, μία, μία, μία, μία κερκόπορτα από την οποία να γίνονται προσλήψεις ε, με, με κάποιο είδους ε, απεμπόληση δικαιωμάτων και με τρόπους αμφίβολους νομικά. Οπότε ε, τελικά να, να, να, κάνουμε κάποιους ορισμούς, κάποιους στενούς, περιοριστικούς και όλα αυτά που θα τα εξετάσουμε. Όμως πρόκειται βεβαίως και για ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να συνεχίσει να μας απασχολεί και μιλώ τώρα για τον τομέα των κατασκευών της οικοδομής. Διότι σε σχέση με αυτό το θέμα ε, πρέπει να, να, να αναγνωρίσουμε ότι ο κλάδος αυτός είναι κάτι σαν το Far West. Ε, έχω ακούσει όλους τους ε, ενδιαφερόμενους, τους και εργαζόμενους και εργοδότες και έχω διαπιστώσει ότι ομόφωνα, ομόφωνα λένε και προτείνουν ότι δεν θέλουν να καλυφθούν από την οδηγία. Δεν θέλουν να είναι στο, στο περιφαρμογή τη, γιατί θεωρούν ότι έτσι, αντί να του λύσει τα προβλήματά του, θα του τα αυξήσει. Αυτό επομένω που θέλω εγώ να πω ότι σκέφτηκα είναι ότι όσον αφορά τι κατασκευέ να μην τι περιλάβουμε στην την οδηγία. Βεβαίω, και επί τη αρχή αυτό δεν είναι τόσο θετικό, δεν είναι καλό να εξαιρούμε κλάδου από τι ρυθμίσει. Όμω, όπω προείπα συμφωνούν όλοι και οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι. Τέλος πάντων, νομίζω και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε κάποιο συμβασμό. Και αυτό το οποίο τελικά είναι σημαντικό και επ' αυτού νομίζω ότι στην Επιτροπή Αποσχόλησης υπάρχει συνένεση, είναι ότι βασική έννοια της οδηγίας είναι η αρχή της ίσης, της ισότιμης μεταχείρισης. Δηλαδή, πιο κατανοητά, τι πάει να πει η ισότιμη μεταχείριση, ότι δηλαδή θα πρέπει στην ίδια χώρα, για την ίδια δουλειά, θα πρέπει οι, τα, τα, τα, φυσικά πρόσωπα να αμείβονται το ίδιο. Τώρα, όσον αφορά τις ε, λεπτομέρειες της εφαρμογής της αρχής, βεβαίω και υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία τα, τα, επεσήμανε ο κύριος Γιακολίνη, τα θέματα κοινωνικής πρόνοιας, ασφάλισης, ε, ε, τα συντεξιδοτικά, Βεβαίως και όλα αυτά είναι περίπλοκα και θα ήταν πάρα πολύ αξιόλογο εάν θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι και να μπορέσουμε να βάλουμε στο κείμενο αυτά τα οποία θέλουμε. Γι' αυτό σας λέω. Τα συζητήσαμε στην Επιτροπή. Οι συγητές, σκιώδει συγητέ και άλλοι και συζητήσαμε, λέγω, την σχέση των διαφορετικών ενιών και των ε, ορισμών που περιέχονται ει αυτή την οδηγία και ει άλλες οδηγίες, ούτω ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση. Και μιλώ τώρα για την ε, οδηγία που αφορά την ενιαία άδεια. Single permit στα αγγλικά. Έχουμε βέβαια και τις διμερείς συμφωνίες. Υπάρχουν διμερείς συμφωνίες μεταξύ ΕΕ και τριών χωρών. Για να δούμε τι θα γίνει με αυτές. Πού θα δοθεί η προτεραιότητα, τι θα κατησχίσει. Να δούμε αν θα πρετανεύσει το κοινωτικό δίκαιο. Όμως αυτό που δεν θα πρέπει να ξεχνούμε είναι το ότι θα πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην νομοθεσία. Θα πρέπει να υπάρχει και σαφήνεια. Όσο γίνεται περισσότερο. Όμως επ' αυτού θα θέλαμε να μας μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. ποια είναι η σχέση μεταξύ κοινοτική νομοθεσίας και διμερών συμφωνιών. Γενικά πάντως θεωρώ ότι είναι κάτι το καλό. Είναι κάτι θετικό. Αυτό το οποίο προσπαθούμε και νομίζω ότι θα βοηθήσει και στην ανταγωνιστικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Έξι είναι οι συνάδελφοι που θέλουν να πάρουν το λόγο. Κυρκόπ, Μπίντσεβιν Τούτε, Σαρτζεντίνη, Μπρόντς και Ο κύριος Κίρκοπ έχει πρώτος το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον κύριο Ιακολίνο για την εργασία του, και να τον ευχαριστήσω για την πολύ επικοδομητική και λογική προσέγγιση που έχει στο ζήτημα και προφανώς συμφωνώ με τα περισσότερα από τα όσα προτείνει. Πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια θετική προσέγγιση, δηλαδή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις να βρούνε το κατάλληλο προσωπικό, κατάλληλο για τους στόχους τους βέβαια, και νομίζω ότι τον έχουμε ένα πιο ευθυγραμμισμένο πλαίσιο για την ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση θα είναι θετικό όχι μόνο για τα άτομα αυτά καθ' αυτά και τις επιχειρήσεις αλλά και για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα για το οποίο έχω κάποιες αμφιβολίες. Το ζήτημα των χρονικών περιόδων και των απαιτήσεων όσον αφορά τα προσόντα και την εμπειρία. Πρώτος εγώ θα είμαι αυτός ο οποίος θα έλεγε ότι προφανώς χρειαζόμαστε προσόντα, είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό και προφανώς θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τους εργαζόμενους να αυξάνουν τα προσόντα τους, ιδίως στις νέες τεχνολογίες. Ωστόσο, κυρία Πρόεδρε, υπάρχουν πολλοί νέοι ταλαντούχοι οι οποίοι εργάζονται στα πλαίσια της πληροφορικής, της επιστήμης και των μαθηματικών και αναφέρω απλώς δύο-τρεις τομείς αυτή τη στιγμή παραδειγματικά. Νέοι λοιπόν οι οποίοι μπορεί ακόμα να βρίσκονται σε φάση απόκτησης των προσόντων τους και οι οποίοι κατά την άποψή μου πρέπει να έχουν και τις απαραίτητες ευκαιρίες. Δηλαδή να μην ε, περιοριστούν εξαιτία των χρονικών αυτών περιόδων που προβλέπονται. Καταρχάς να δείξουμε εμπιστοσύνη σε επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν μόνος να αποφασίσουν την θετικό για αυτές. Και επίσης η βιωσιμότητα, η μακροζωία των υπηρεσιών, της υπηρεσίας, η αρχαιότητα ουσιαστικά δεν σε κάνει απαραίτητα τον καλύτερο υποψήφιο. Το έχω δει και εγώ ίδιος αυτό στα πλαίσια τόσο του επιχειρηματικού μου βίου όσο και στα πλαίσια της εντολής μου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επομένω πιστεύω ότι θα πρέπει να ενθαρρύνουμε ιδιαίτερα τους νέους και να προσλάβουμε ουσιαστικά περισσότερους νέους, ιδίως όσον αφορά τον τομέα των νέων τεχνολογιών. Οτιδήποτε μας αποσπά από το στόχο αυτό πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το επανεξετάσουμε. Για όλα τα υπόλοιπα συγχαρητήρια στον κύριο Ιακολίνο. Σας ευχαριστούμε κύριε Κυρικόπη, κυρία Μπλενταβιτούτιν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Γιακολίνο για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Και εξάλλου δεν είναι καινούριο αυτό. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις σε σχέση με την έκθεση αυτή και υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία καταρθώσαμε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις. Ελπίζω ότι θα τύχουν υποστήριξη και από την Επιτροπή τα σημεία στα οποία εμείς καταλήξαμε σε κάποια συμφωνία. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που συζητήσαμε και την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Η τροπολογία 19 που αφορά την ίση μεταχείριση των φύλων ε, δυνατότητα συμφιλίωσης ε, οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, κυρίως για τις γυναίκες, ούτως ώστε να υπάρχουν καλύτερες ευκαιρίες ένταξης στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μια τροπολογία του κυρίου Γιακολίνο και προτείνεται να καθορίζουν τα κράτη-μέλη τις συγκεκριμένες διατάξεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εγώ βλέπω ότι θα υπάρχει δυνατότητα πολλών και διαφορετικών συνθήκων ανάλογα με την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος και δεν θα δίνουμε τη δυνατότητα ε, ίσης μεταχείρισης. Εδώ ελπίζω ότι θα υπάρξει κάποια δυνατότητα ε, συμβιβαστικής τροπολογίας και για την άδεια εργασίας εργαζομένων από τρίτες χώρες Συμφωνώ με την προτινόμενη λύση η οποία συμβάλλει προς την επανένωση των οικογενειών. θα πρέπει να συμφωνήσουμε ε, για το σύστημα που θα ισχύσει σχετικά με την ε, μετάθεση ενός εργαζομένου από τρίτη χώρα ε, ενός εργαζομένου που είναι υπήκος τρίτης χώρας από το ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλο. θα πρέπει να ισχύουν οι ίδιες συνθήκες εργασίας και οι ίδιες μισθολογικές συνθήκες. Ακούσαμε και από τον εισηγητή αλλά και από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου και της Επιτροπής ότι είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε κοινού ορισμούς και οι ορισμοί θα πρέπει να είναι ούτε πολύ ευέλικτοι ούτε πολύ περιοριστικοί. Θα πρέπει να μας δίνουν τη δυνατότητα σωστής κατανόησης. Θα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι εννοούμε όταν χρησιμοποιούμε κάποιο όρο να ξέρουμε τι εννοούμε όταν λέμε διοικητικά στελέχη ή ασκούμενοι πτυχιούχοι ή ειδικευμένοι υπάλληλοι. Και έχουμε κάνει συγκεκριμένες προτάσεις στις τροπολογίες μας σχετικά με τους ορισμούς. Παραδείγματος χάρη για τα διοικητικά στελέχη. Υπάρχει μια συγκεκριμένη τροπολογία για τις συνθήκες εργασίας και για τις ε, μισθολογικές συνθήκες. Επίσης για τις περιόδους, για χρονικές περιόδους που προβλέπονται για τους ε, μετατιθέμενους από τρίτες χώρες προτείνεται μια περίοδος εννέα μηνών αλλά συζητείται και μια περίοδος μηνών ή μηνών ή 12 μηνών. Η δωδεκα μηνων πάντοτε έχει σημασία Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ε, συμφωνία, γιατί το έγγραφο σε γενικές γραμμές ε, είναι σωστό. Και ε, κάτι ακόμη σε σχέση με αυτό που είπε η κυρία Γιάκον Σάρη για τον τομέα των κατασκευών, Εδώ θα ήθελα να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Αυτά από δική μου πλευράς. Πάντως γενικά το κείμενο είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. λέει η κυρία Βίξτρομ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Σαλβατόρα Γιακολίνο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει για το θέμα αυτό. Είναι σημαντικό αυτό το θέμα, ε, διότι η παγκοσμιοποίηση απαιτεί κινητικότητα. Ε, πρέπει και εμείς να επιτρέπουμε ε, στους πολίτες να μετακινούνται, να εργάζονται και να οργανώνουν τη ζωή τους σε άλλο τόπο σε σχέση με τον τόπο γέννησής τους. Είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις ε, να υπάρχουν αυτές οι διατάξεις. Δύο περιοριστικοί ορισμοί είναι απαραίτητοι για να μην υπάρχουν περαιτέρω κατηγορίες σε αυτήν την οδηγία και επίσης συμφωνούμε να συνοδεύονται οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι από τις οικογένειές τους, διότι υποστηρίζουμε την επανένωση των οικογενειών και την συμφιλίωση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Αυτό ισχύει και για αυτήν την οδηγία και σε άλλες οδηγίες και άλλα κείμενα που έχουμε επεξεργαστεί. Ελπίζω ότι θα εγκρίνουμε ένα συνολικό πακέτο για την νόμιμη μετανάστευση. Η θέση του κυρίου Γιακολίνου είναι θετική και ελπίζω ότι ότι θα μπορέσουμε σύντομα να εγκρίνουμε αυτό το κείμενο, διότι τα θέματα της ενδοεπιχειρησιακής μετάθεσης ε, για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντικά και πέραν της οικονομικής κρίσης που αυτή τη στιγμή ζούμε στην Ευρώπη. Πρέπει να έχουμε ένα όραμα για το μέλλον και να χρησιμοποιούμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είναι οι ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις, για να επιτύχουμε το στόχο της ευημερίας και της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Βίξτον, κυρία Σαρτζεντίνη. Um, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιακολίνο, διότι κατάφερε να καταλήξει σε κάποιες συμβεστικές λύσεις, οι οποίες, από ό,τι φαίνεται, τους περισσότερους εξημών τους ε, καλύπτει. Τουλάχιστον εμένα, περισσότερο το το λέει. Έχω κάποιες ε, μικρές παρατηρήσεις πάντως. Και ήδη έχω πει ότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο το τι ποινέ θα θεσπιστούν για τους εργοδότες και εάν θέλουμε να τηρούν τη διατάξη του εργατικού δικαίου ή για τη μετανάστευση θα πρέπει οι εργοδότες να ξέρουν τι επιτρέπεται γιατί απαγορεύεται. Κυρίως εμείς μιλούμε για τις κυρώσεις που αφορούν τους εργαζόμενους και τους μετανάστες. Άρα θα πρέπει με προσοχή να δούμε τι ισχύει για τους εργοδότες, τι κυρώσεις προβλέπονται. Επίσης, έχετε ενσωματώσει αυτά τα οποία είχαμε προτείνει στις ε, τροπολογίες, ε, τις συμβαστικές, ας πούμε στην υπαριθμό 15. Τώρα έχω κάποια άλλη πρόταση που θα ήθελα να σας αναφέρω, ότι δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα της ε, διακριτικής ευχαίρεσης όσον αφορά αυτές τις κυρώσεις. λέει δυνατόν να έχουν ε, αυτές τις ε, διαδικασίες κλπ. κλπ. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει αυτό να το κάνουμε σαν υποχρεωτική ρύθμιση. Να μην λέει may, να λέει shall το αγγλικό κείμενο. Όχι δυνατή, αλλά θα θεσπίσουν κάτι. Θα κάνουν. Θα πρέπει επομένω να γνωρίζουν και οι εργοδότε το τι γίνεται. Τι γίνεται για αυτού του εργαζόμενου οι οποίοι θα δουλεύουν δίπλα-δίπλα και θα είναι από διαφορετική χώρα και να ξέρουν ότι θα πρέπει να τη χάνουν οι μεταχείριση αυτοί οι εργαζόμενοι. Τώρα, εδώ αναφέρεται πώς και από ποιους όρους δίνεται, δεν δίνεται η άδεια, η έγκριση και λέτε για το θέμα της ποσότητας των αδειών του αριθμού. Ε, κοιτάξτε, ε, αυτό ισχύει έτσι κι αλλιώς αλλά αυτοί εδώ είναι, κινούνται στις, στα πλαίσια της ίδιας εταιρεία. είναι εδώ δεν παίρνουν τη θέση κανένας. Από τρίτη χώρα έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, όσον αφορά τους πράσινους, ο αριθμός δεν θα πρέπει να λαμβάνεται ως κριτήριο για αυτές τις ε, ενδοεπιχειρησιακές ε, μετακινήσεις. Τώρα, τελευταίο θέμα. Έχω ένα ερώτημα για τη δεύτερη τροπολογία. Εκεί που περιλαμβάνεται ένα νέο σημείο όσον αφορά το κεφάλαιο κάποιων εταιριών σε σχέση με με το μετοχικό κεφάλαιο και, του, και τις, τις, ψήφους που οι μετοχές δίνουν στους μετόχους. Θέλω να διευκρινιστεί αυτό, δεν καταλαβαίνω δηλαδή το πολιτικό ελαττήριο για μια τέτοια ρύθμιση. Τώρα, τελευταίο, θα ήθελα επ' αυτού να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη γνώμη της για αυτό το οποίο είπα όσον αφορά το κριτήριο του αριθμού των μεταναστών ή του αριθμού τη έγκριση εισόδου των μεταναστών, να μου πει αν αυτό ε, μπορεί εδώ πέρα να το επικαλεστεί κανεί για αυτόν τον κανονισμό. Ευχαριστούμε κύριε Σαντζεντίνη, κύριο Μπλάντ. Ευχαριστώ. Οι επικριτέ του καπιταλισμού Πολλέ φορέ κάνουν έτσι γελιογραφίε για την ε, κακομεταχείριση των εργαζόμενων σαν να ήταν αντικείμενα, σαν να ήταν μέσα παραγωγή. Όταν εδώ τώρα, τώρα που μιλάμε για αυτού ε, του, του, τους συγκεκριμένους εργαζομένους και για του ανθρώπινους ε, ανθρώπινους πόρους. Ε, έτσι δικαιώνομαι αυτού του επικριτέ του καπιταλισμού, του γερογράφους. Βεβαίω και πρόκειται για ανθρώπινα όντα. Δεν μιλούμε εδώ για πόρους, ανθρώπινους πόρου. Οπότε, αυτή η οδηγία ICT, είδατε, ω και εγώ κάθομαι και το λέω, ε, το λέμε κάτι σαν απόσπαση, σαν μετάθεση και αυτό όμως βοηθάει και τα μέλη τη οικογένεια. Ε, οπότε για μένα είναι ένας τρόπος να υπάρχει διευκόλυνση, όχι ε, κάποιο είδους μετάθεση, απόσπαση ε, προσωρινή, αλλά αυτό είναι κάτι σαν Ε, παραμονή. Επομένως εδώ πέρα μας καρεύεται μια, μια μετανάστευση ανεξέλεγκτη. Όποιος έρχεται εδώ θα μείνει. Και επομένως σε σχέση με τις εταιρείε, αυτό το οποίο τώρα βλέπουμε είναι ότι κάποιες πολυεθνικές να μας υπαγορεύουν τι νομοθετήματα πρέπει να θεσπίσουμε τόσο ώστε να, μπορέσουμε να, να, να παρακάμψουμε το, το δίκαιο για τους ελέγχους της μετανάστευσης και να τη διευκολύνουμε. Γιατί χρειάζεται μετανάστευση. Μας λέει αυτό το έγγραφο και το λένε και άλλοι, βοηθάει γιατί το χρειάζονται επιχειρήσεις και εταιρείε και ότι οι άνθρωποι υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο για να εξυπηρετούν τις εταιρείε. Παραδόξω για το δω και δικαιώνει και η αριστερά τις πολυεθνικές. Η μετανάστευση έχει σημαντικές συνέπειες για πολλές χώρες και οι ψηφοφόροι μας ανησυχούν και βεβαίως και για το αν θα χάσουν τη δουλειά τους, αλλά θα πρέπει όλα αυτά να τα πάμε στην άκρη γιατί το ζητά η παγκοσμιοποίηση. Και οι τη παγκοσμιοποίηση λένε ότι θα πρέπει επομένω, σαν πρόκειται για πιόνια σκακιού, να πάνε πέρα δόθε όπου βολεύει οι εργαζόμενοι, και οι πολιτικοί, οι πολιτικάντες τέλο πάντων για αυτοί στρατεύονται στο, στο σκοπό της παγκοσμιοποίησης για να την εξυπηρετήσουν. Ευχαριστούμε. Κύριε, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν νομίζω θα πρέπει να ανησυχείτε γι' αυτό. σε ένα σημείο. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε περί τίνος πρόκειται. Θέλουμε να διευκολύνουμε τις ενδοεπιχειρησιακές μεταθέσεις. Θέλουμε να το κάνουμε περισσότερο ελκυστικό, διότι έχει σχέση με την ανταγωνιστικότητα, με την ίση μεταχείριση. Και θέλουμε να κάνουμε και κάτι ρεαλιστικό και πρακτικό τελικά. Αυτή είναι η βασική μας ε, φιλοσοφία, αυτό είναι το σκεπτικό μα και δεν πρέπει να ξεχνάμε το σκεπτικό μα σε αυτά τα οποία κάνουμε στην πράξη. Κάποιες παρατηρήσεις τώρα. Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, δουλειά που έχει κάνει και για την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε, ούτως ώστε να καταλήξουμε σε κάποια σημεία σημαντικά ε, για όλους μας, ε, τα οποία τα βλέπουμε τώρα στην έκθεση. δεν θα μπορούσαμε να βρούμε ε, ε, ε, κάποια τέλεια λύση για τους ορισμούς. Ο όρος trainee, ο όρος του ασκούμενου με βρίσκει τελικά σύμφωνη, αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξουμε τελικά σε ορισμούς αποδεκτούς. Και σε σχέση με τη δική μου χώρα υπάρχουν αρκετά προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή και τη χρήση των ορισμών. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι σημαντικό είναι η χρονική περίοδος, οι εννέα μήνες που αναφέρονται για παράδειγμα. Πάντοτε δημιουργούν προβλήματα. Και το, η τροπολογία 8 στο άρθρο 3 3Γ, 3 3G μάλλον, δεν ξέρω αν βασίζονται τα τρία χρόνια τα οποία εκεί αναφέρονται. Επίσης, ε, σαν συμβιβαστική λύση, από 12 μήνες κατεβήκαμε στους 9 μήνες για ε, την απαιτούμενη πείρα. Δεν ξέρω και αυτό αν είναι σωστό το να έχουμε τέτοιους περιορισμούς. Θετικό είναι το ότι υπάρχουν κυρώσεις και έλεγχοι. Είναι σημαντικό να υπάρχουν επιθεωρήσεις. Νομίζω η κυρία Σαρζεντίνη είπε ότι πρέπει να γίνονται έλεγχοι και επιθεωρήσεις και εγώ συμφωνώ με αυτό. Πιστεύω ότι η ιδέα είναι σωστή και θα πρέπει και να εμφανίζεται στο κείμενο ακόμη περισσότερο. Όσον αφορά την ίση μεταχείριση, ε, εδώ πρέπει να το τονίσουμε περισσότερο από ό,τι στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων. Και αυτό ισχύει και για τις αποδοχές. Η κυρία Μπλίνκεβιτσούτε και η κυρία Θερτζεντίνη προσπάθησαν ε, να κάνουν κάποια πρόταση για το νέο άρθρο 16 και για το 15α. Εδώ χρειαζόμαστε πιο ξεκάθαρες διατυπώσεις για την ίση μεταχείριση στο χώρο εργασίας και θα πρέπει να ισχύουν αυτά τα οποία ισχύουν ε, στο κάθε κράτος μέλος και στις συλλογικές συμβάσεις. Για την επανένωση των οικογενειών βρίσκω θετικό το ότι προτείνεται ένα τέτοιο μέτρο. Αλλά πρέπει γενικά να το σκεφτούμε κατά πόσο είμαστε πολύ γενναιόδοροι στα μέτρα επανένωσης των οικογενειών. Όταν μιλάμε για ανταγωνισμό, θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε αυτές τις χώρες θα πρέπει να έχουν και κάποια κίνητρα, να ξέρουν ότι αν πάω θα έρθει και η οικογένειά μου χωρίς να έχω τεράστια προβλήματα για την επανένωση της οικογένειας. Γι' αυτό λοιπόν ας δούμε το κατά πόσο είμαστε γενναιόδοροι στην επανένωση των οικογενειών. Για τις κυρώσεις ε, καλή είναι η διατύπωση και αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Έρνστ και πριν επανέλθω στον εισηγητή, θέλω να ζητήσω από την Επιτροπή να απαντήσει στην ερώτηση της κυρίας Γιακονσάρη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως σας είπα και χθες στην Επιτροπή Απασχόλησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρότεινε να ασχοληθούμε με το ζήτημα της εφαρμόσιμης νομοθεσίας όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση. Θεωρώ όμω ότι εδώ πέρα αναφερόμαστε περισσότερο στο σύνδεσμο που υπάρχει με τις διμερείς συμβάσεις, τις οποίες μπορεί να προβλέπεται ότι όσον αφορά την κοινωνική ασφάλιση, η ασφάλιση της χώρας προέλευσης μπορεί να διατηρηθεί Όσον αφορά το βασικό σκεπτικό και το, τα όσα προτείνονται, ουσιαστικά οι διμερείς συμφωνίες θα μπορούν να ισχύουν αν προβλέπουν πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Από ό,τι κατάλαβα αυτή είναι η βασική σας ιδέα, το βασικό σας σκεπτικό. Αυτό είναι ενδιαφέρον βέβαια, ενδεχομένως να μπορούσαμε όμως να το εξετάσουμε με μεγαλύτερες λεπτομέρειες. Πάντω δεν περιέχεται στην πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα φαίνεται ενδιαφέρουσα πρότασή σα και θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε περαιτέρω να επανέλθω και σε κάποια άλλα ζητήματα όσον αφορά την ποσότητα, τον όγκο. Προφανώς τα κράτη-μέλη είναι τα πλέον αρμόδια να αποφασίσουν ποια θα είναι η δυνατότητα εισδοχής ξένων υπηκών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τη χώρα τους. Αποφασίζοντας βέβαια γι' αυτό, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν τις διεθνείς συμβάσεις για το εμπόριο. Τέλος, ένα ζήτημα το οποίο θίξαμε πριν από λίγο, η επαγγελματική εμπειρία. Ζήτημα το οποίο επανέρχεται και στις συμβαστικές τροπολογίες. Ουσιαστικά έχουμε ένα αίτημα για μία πενταετή επαγγελματική εμπειρία και αυτό δεχομένω να αποκλείει κάποιους νέους ανθρώπους, ιδίως στον τομέα της πληροφορικής. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να εξετάσουμε λίγο περισσότερο και αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Σμίτ. Δίνω και πάλι το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Ιακολίνο. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ πρόεδρε. Άκουσα όλες αυτές τις παρεμβάσεις από τους συναδέλφους. Άκουσα την κυρία Μπλικαμβιτσούτε, την κυρία Γιάκον Σάρη, την κυρία Σαρτζεντίνη, τον κύριο Μπρόνσα, την κυρία Έρνστε. πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι έχουν κάνει πολύ λογικές, ε, πολύ ε, κέρυες προτάσεις, τις οποίες θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω στην ε, έκθεση αυτή. Το είπα ήδη και το ξαναλέω και τώρα, ότι ο κατασκευαστικός τομέας δεν περιλαμβάνεται στην πρόταση. Προσπαθούμε παρόλα αυτά να έχουμε ένα ευρύ πεδίο εφαρμογή στι διαπραγματεύσει τι οποίες διεξάγουμε. Συναντήθηκα επίσης με ομάδες που εκπροσωπούν εργοδότες και εργαζόμενους. Προφανώ οι απόψει διήστανται, είναι διαφορετικές πολλέ φορές. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ε, αν θέλουμε να έχουμε μία ευρεία εφαρμογή της οδηγίας για την ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση, δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε τον κατασκευαστικό τομέα. Διότι πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό τομέα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και έναν τομέα που περιλαμβάνει πολύ μεγάλες ροές εργαζομένων και πολλές φορές για σύντομα βέβαια χρονικά διαστήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο τομέας αυτός. Δεν νομίζω λοιπόν θα πρέπει να εξαιρεθεί ο τομέας αυτός. Το λέω με σαφήνεια αυτή τη φορά. Μπορεί να μην έγινε κατανοητός πριν από λίγο. Προφανώς θα πρέπει να έχουμε ισότιμη μεταχείριση όσον αφορά τους εργαζομένους και προφανώς θα πρέπει να προβλέπεται και ασφαλιστική κάλυψη και βέβαια και οι αντίστοιχες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Ως προς το ζήτημα αυτό θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις απαραίτητες επαφές με τις χώρες προέλευσης και ότι θα πρέπει να προβλέπονται απαραίτητε συμφωνίε, πολλέ φορέ ακόμα και διμερεί συμφωνίε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι ε, η κοινωνική ασφάλιση του αποσπασμένου εργαζομένου θα συνεχίσει να ισχύει και στην ε, χώρα στην οποία πηγαίνει. Θέλουμε να καταλήξουμε προφανώ εμεί σε έναν εναρμονισμένο κανονισμό που θα αποφεύγει την, το κατακρεματισμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις διαφορετικές διμερείς συμφωνίες. Και βέβαια να υποστηρίξουμε και τους νέους. Ο κύριος Κίρκοπ το είπε ότι θα πρέπει να δώσουμε τόπο στα νιάτα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να προβλέπετε ένα ελάχιστο επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας, το οποίο όμως δεν θα αποκλείει από τα νομοθετήματα αυτά τους νέους. Αναφερόμαστε λοιπόν σε νέους οι οποίοι έχουν ήδη μια σύμβαση με μια εταιρεία, είναι ήδη μέρη, μέλη του συστήματος και τους δίνουμε εδώ πέρα τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν περισσότερο την επαγγελματική του ζωή, να εργαστούν για ένα άλλο τμήμα της ίδιας εταιρεία σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία Μπλικενβιτσούτε μας είπε ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη πρόσβαση ακόμα και στους συζύγους ή τις συζύγους. Καταλαβαίνετε βέβαια ότι ο ICT, ο υφιστάμενος ενδοεπιχειρησιακή μετάθεση, δεν είναι απαραίτητα άντρα, μπορεί να είναι και γυναίκα. Και προφανώς θα πρέπει να καλύψουμε και του τις συζύγους. Αν κάποιος μετατίθεται για παράδειγμα από τη Γαλλία στη Δανία, από την Μάλτα στην Κύπρο, δεν μπορούμε να πούμε στον αποσπασμένο αυτό εργαζόμενο ότι ο η σύζυγός σου θα πρέπει υποχρεωτικά να βρει εργασία στην χώρα υποδοχής δεν μπορεί αυτό να αποτελεί δηλαδή απέτησή μας, απόλυτη απέτησή μας. Και να έχουμε εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούμε να τους αποτρέψουμε από το να φέρουν μαζί τον ή τη σύζυγό τους. Αυτό θα ήταν αρνητική διακριτική μεταχείριση. Είναι πολύ σημαντικό να μπορεί όλη η οικογένεια να μετακομίζει και πιστεύω ότι όντως στην παράγραφο 20 το ΜΕΙ μπορεί να γίνει ΣΑΛ, να λέγεται δηλαδή ξεκάθαρα ότι τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν για τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην αγορά εργασίας για την σύζυγο ή τον σύζυγο του υφιστάμενου ενδοπεχειρησιακή μετάθεση του αποσπασμένου. Και συμφωνώ επίση με την πρόταση η οποία ακούστηκε πριν από λίγο ότι θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να έχει και ένα κάποιο βαθμό ευελιξία προκειμένου να μπορεί να προσαρμοστεί το σύστημα αυτό. Δεν νομίζω ότι σε περίοδο, ιδίω σε περίοδο οικονομική κρίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα δίσκαμπτο. Πρέπει επίσης να εργαστούμε περισσότερο για την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα του συστήματος εν γέννη. Συμφωνώ επίση με την κυρία Σαρτζεντίνη όσον αφορά το ζήτημα των κυρώσεων. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα ευαίσθητο και λεπτό ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο το συζητήσαμε πολλές φορές στο παρελθόν και προβλέπονται επιπλέον κάποιες προϋποθέσεις αυτή τη στιγμή σε σχέση με το προϋπάρχον κείμενο όσον αφορά τον όγκο των εισρών της εισδοχής προς τις τρίτες χώρες και μπορούμε εδώ πέρα να αφαιρθούμε και στο άρθρο 79 παράγραφος 5 όπου περιγράφεται μια γενικότερη αρχή για την ε, επανεισδοχή και για τις ε, ροές εργαζομένων από τη μία χώρα στην άλλη. Δεν νομίζω λοιπόν όμως ότι οι εργαζόμενοι από τις τρίτες χώρες θα πρέπει να, ο αριθμό τους να είναι δυσανάλογο σε σχέση με τον αριθμό των υπόλοιπων εργαζομένων που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να σας πω επίσης, σε σχέση με μια άλλη παρατήρηση που έγινε, ότι ορισμένες από τις διατάξεις που βλέπετε εδώ πέρα έχουν ε, διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να συνάδουν με τις συμβάσεις που ισχύουν αυτή τη στιγμή στην αγορά εργασίας. Επομένως, ακούγοντας τις δικές σας προτάσεις, κάναμε τις αντίστοιχες προτάσεις για τις πληρωμές, αποδοχές, για την πενταετή περίοδο, Υπάρχει μάλιστα η ε, συμβαστική τροπολογία 4 που ασχολείται με την περίοδο αυτή και προσπαθούμε να διευθετήσουμε και το ζήτημα της επαγγελματικής εμπειρίας στην ίδια τροπολογία. Χρησιμοποιούμε εδώ πέρα μία διάταξη η οποία ισχύει και για την οδηγία για την μπλε κάρτα, την οποία έχουμε εγκρίνει ήδη στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βέβαια μπορούμε να το εξετάσουμε περαιτέρω το ζήτημα αυτό εφόσον δεν συμφωνείτε με την υφιστάμενη διατύπωση. Νομίζω ότι οι ελάχιστες προϋποθέσεις ε, εισόδου μάλλον θα πρέπει να περιοριστούν και όχι να επεκταθούν κατά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Αναφερθήκαμε στις οικογένειες, στην επανένωση οικογενειών, και ακόμα και στους ορισμούς προσπάθησα να πετύχω την κατάλληλη ισορροπία, δηλαδή να μην είμαι αρκετά περιοριστικός στους ορισμούς και από την άλλη όμως να μην αφήσω τα πράγματα πάρα πολύ ανοιχτά όσον αφορά την ερμηνεία των διαφόρων ορισμών. Ως προς το πεδίο εφαρμογή επίσης της οδηγίας πάλι πρότεινα μια πιο ισοσκελισμένη προσέγγιση. Αναφέρομαι και στα διοικητικά στελέχη και τους διοικητμένους υπαλλήλους αλλά και στους ασκούμενους πτυχιούχους. Αναφερόμενος στα διοικητικά στελέχη, αναφέρομαι και σε επιμέρους πτυχές ε, της ε, θέσης τους, ότι μπορεί να έχουν κάποια συγκεκριμένα καθήκοντα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, ότι πρέπει να πετύχουν κάποιους συγκεκριμένους μετρήσιμου, μετρήσιμους στόχους. Άκουσε επίσης και τόσο είπε ο κύριος Μπρόνς και θα ήθελα να, τον, να του πω ότι η οδηγία αυτή σε καμία περίπτωση δεν, δεν αποτελεί έναν τρόπο να αποφύγουμε ή να μην συμμορφωθούμε με τους κανόνες για την νόμιμη μετανάστευση. Προσπαθήσαμε απλώς σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα να θεσπίσουμε μία οδηγία η οποία θα διευθετεί καλύτερα τις ροές της νόμιμης μετανάστευσης με βάση τις ανάγκες αγοράς εργασίας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν άλλα κρεμή ζητήματα αυτή τη στιγμή ή άλλα ερωτήματα εκ μέρου σα. Προφανώ όμω, αν υπάρχουν κάποια κρεμή ακόμα ζητήματα, θα τα διαπραγματευτούμε μαζί. Θέλουμε να ρυθμίσουμε τι μεταναστευτικέ ροέ και θέλουμε ουσιαστικά να αντικατοπτρίζονται στι ανάγκε αγορά εργασία. Μιλήσαμε για την ισότιμη μεταχείριση. Συμφωνούμε νομίζω όλοι ότι θα πρέπει να προβλέπονται συγκεκριμένε κυρώσει. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε δυνατή κάθε πιθανή, με συγχωρείτε, αρνητική μεταχείριση του συστήματος. Πρέπει επίσης να δούμε τι κάνει και το Συμβούλιο σε σχέση με τη σημαντική αυτή οδηγία και ελπίζω ότι θα έχουμε κάποια θετικά νέα από το Συμβούλιο όσον αφορά την, κινητικότητα των εργαζομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το οποίο θέλουμε να πετύχουμε εν τέλει είναι να υπάρχει μία αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των εργαζομένων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης κάθε φορά που ε, μετατίθενται οι εργαζόμενοι. Επίσης δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε την τριετή χρονική περίοδο η οποία προβλέπεται στην οδηγία και δεν θέλουμε η χώρα υποδοχή να είναι αυτή η οποία θα πρέπει να υπομειστεί το διοικητικό βάρο αν ένα αποσπασμένο εργαζόμενο τελικά δεν επιστρέψει στην ε, χώρα προέλευσή του. Ελπίζω λοιπόν ότι οι συμβαστικέ τροπολογίε κατάφεραν να καλύψουν όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία έχετε θίξει. Προφανώ όλα μπορούν να τροποποιηθούν ακόμα περισσότερο εφόσον το επιθυμείτε. Θα έχουμε και άλλε συνεδριάσει και ελπίζω ότι στι 25 Ιανουαρίου θα έχουμε καταλήξει πλέον σε ένα κείμενο το οποίο θα χαίρει πολύ μεγάλη υποστήριξη. Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τους ορισμούς, ελπίζω θα καταφέρουμε να έχουμε μία ενιαία προσέγγιση προκειμένου να βελτιώσουμε τη συνεργασία ανάμεσα στη δική μας Επιτροπή και την Επιτροπή Απασχόλησης και ελπίζω ότι τελικά στην τελική ευθεία θα καταφέρουμε να πετύχουμε τους κοινούς μας στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Ιακολίνο, λέει Πρόεδρος. Σας υπενθυμίζω ότι τον Ιανουάριο θα επανεσυζητήσουμε την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ενεργή συμμετοχή τους. Το επόμενο σημείο στη μερίσια διάταξη είναι οι ψηφοφορίες μας. Θα ξεκινήσουμε στις 11.45 ακριβώς με τις ψηφοφορίες. Έχετε λοιπόν 3-4 λεπτά ακόμη. Okay, colleagues, let's uh, Συνάδελφοι, ας ε, συνεχίσουμε τις εργασίες μας και αρχίζουμε τις ψηφοφορίες, λέει η Πρόεδρος. Έχουμε για να, να ψηφίσουμε τρεις εκθέσεις. Η πρώτη είναι το σχέδιο κανονισμού Κοινοβουλίου σε σχέση με την τροποποίηση του οικονομισμού 1931 του 2006 για την συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνιγκρατ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή. Δεν έχουμε τροπολογίες για αυτή την έκθεση. Οπότε ψηφίζουμε. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Σαφώς και εγκρίνεται. Χρειαζόμαστε ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τελική ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες, συνάδελφοι. Όχι. Και κύριε Σαρτζεντίνη. Να δούμε τι θα κάνει. Ψηφίζουμε πέρας. Ομοφόνος εγκρίνεται. Α, έχουμε μία αποχή. Επόμενη. Το σχέδιο της εκθέσεως και Επιτροπή όσον αφορά την ε, πρόσβαση του κοινού ή το δικαίωμα ενημέρωση μάλλον στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Συγχαρητήρια στην κυρία Σίπελ που έφτασε μέχρι εδώ, αλλά και τους του ε, σκιώδους ηγητές γιατί ήταν σκληρές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για να επιτευχθεί συμφωνία. Τώρα, πριν προχωρήσουμε στην ε, ψήφιση, σας ε, ανακοινώνω ότι ε, υπήρξε συμφωνία όλων των σχεδόν εισηγητών, ούτω ώστε να έχουμε το ενιαίο κείμενο, από αυτού να υπάρχει συμφωνία με όλες τις τροποποιήσεις του κειμένου και ψηφίζουμε τώρα 145. Ψηφίζουμε, ψηφίζουμε ε, εδώ πέρα όλες μαζί είναι υπέρ, τι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται, είναι σαφές και τώρα θα κάνουμε για το ψήφισμα μια ηλεκτρονική ψηφορία. Πέρας. περας ψηφορία. ψηφορίας. 46-2. Με δύο εποχέ. Όχι, δύο υπέρ, δύο υπέρ διαφωνεί πρώτο. Και τώρα πάμε στο σχέδιο κειμένου που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής. Κύριε Κάσμα, θέλετε το λόγο. Είστε ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Κυρία Γκάλ. Υπάρχει στην λίστα για την ψηφοφορία ένα λάθος. Κοιτάξτε τις σελίδες συνάδελφοι 4 και 5. Εκεί που λέει συμβιβαστική 7. Εάν αυτή εγκριθεί, 102, 103, 104 και 105 αυτές οι τροπολογίες ε, θα πρέπει να καταπέσουν. Ψηφίζουμε λέει πρόεδρος τώρα. Έχουμε δύο. Σαν που δεν έχουν την κάρτα. Θα χρειαστεί η κάρτα μάλλον. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά. αποχές. Εγκρίνεται. Έλεγχος. Έχουν μία παραπάνω ψήφο οι σοσιαλιστές. Πέρασε. 34-16, χωρίς αποχές. Άρα, απορρίπτωτο. Όχι καταπίπτει. Συμβαστική 2, υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 3. 70-24, 72-73-74 ε, υπέρ κατά, αποχές. Θα πρέπει να γίνει έλεγχος, έλεγχος για τη συμβαστική 3. Ψηφίζουμε. Πέρας. 31, 19. 33 είπε ο πρόεδρο, 31 έλεγαν οι ηλεκτρονικοί πίνακες. Πάμε τώρα στη συμβαστική υπερθυμών 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται, αλλά ας κάνουμε έλεγχο. Κύριε Γκάλ. Ίσως να τα κάνουμε όλα ηλεκτρονικά για να ωφεληθούν όλοι, γιατί από ό,τι φαίνεται έχουμε όσο από το πλήστον σαφή αποτελέσματα κάθε φορά υπέρ ή κατά. Μήπως αν τα κάνουμε ηλεκτρονικά είναι καλύτερα για όλους. Ναι, ναι, ναι. Ας το κοιτάξουμε. Όπως είπα, τελεπρόεδρος, οπότε πάμε στο 4 με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίζουμε. 31-18. 33 υπέρ διορθώνει ο πρόεδρος, προφανώς αυτοί που δεν έχουν κάρτα, 33-18. Και πάμε τώρα στην συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. αποχέ Και εγκρίνεται. 27 και 41. Υπέρ. Κατά. αποχέ. Δεν είναι σαφέ θα πρέπει να γίνει έλεγχο. Ψηφίζουμε. Πέρας. 31, 19. Μία εποχή. Παρακαλώ σηκώστε το χέρι γιατί είναι δύσκολο από εδώ να δούμε τι γίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτωτε. Τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπής αναφορών 4. Υπέρ, κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 82. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 84. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 και 86 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 επίσης κατά Καταπίπτει. 87 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβεστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επτά. Συγγνώμη Επτά συμβαστική. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα του 34. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Κατόπιν. 8. Συμφαστική 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν δέκα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέκα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 9 της Επιτροπής Αναφορών υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Αύκο 7 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 126. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 127. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Αύκο. 8. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41. Ήδη ψηφίστηκε με το 27, πάμε τώρα στην αναφορών. 10, καταπίπτει 130, υπέρ. Κατά, από συγκρίνεται. Πρώτα ευχαριστώ. Το συζητήσαμε με τον εισηγητή στην τελευταία φάση όσον αφορά την επομένη, την 131. Έχω μια προφορική τροπολογία για να αντικαταστήσουμε την 200 ε, από την 50. Ε, οπότε ξέρω ο κ. Κάστον συμφωνεί. Ποιοι είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Υπέρ κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα πάμε στην 12 αναφορών. Υπέρ. Λοιπόν, Τώρα θα ψηφίσουμε για την τροπολογία 131, όπως έχει τροποποιηθεί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία Επιτροπής Αναφορών 12, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 42, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με την ίδια πλειοψηφία, 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 134 υπέρ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται Τώρα, τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 53 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα, 54 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1. Όχι, όχι, συγγνώμη, 55 δεν καταπίπτει, 55 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 57. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, συγγνώμη, ξέχασα μία. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, α όχι, 61 καταπίπτει. Τροπολογία 11 υπέρ, κατά, Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται μάλλον 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 66 υπέρ, όχι, καταπίπτει, συγγνώμη, τροπολογία 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 67 καταπίπτει. Και περνάμε, κυρία Ζώνα, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα ε, να κάνω ένα διαδικαστικό αίτημα. Θα ψηφίσει κατά η ομάδα του ΕΛΚ. Αντιπροσωπεύουμε μία μειοψηφία βέβαια. Και γι' αυτό θα κάνουμε μία δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 51.3, μία δήλωση μειοψηφίας και παρακαλούμε να καταχωρηθεί η δήλωσή μας στα πρακτικά. Ευχαριστώ κυρία Ζώμε. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Περιμένω να διαβάσω την δήλωση της μειοψηφία και ευχαριστώ πολύ την κυρία Ζόμερ για αυτό το διαδικαστικό θέμα που ανέφερε και πριν περάσουμε στην τελική ψηφοφορία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την ευρία και δύσκολη ψηφοφορία την οποία πολύ αποτελεσματικά διεκπαιρεώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. The, the vote is closed. ψηφοφορίας. 33 υπέρ, 17 κατά, 2 αποχές. Ευχαριστούμε κύριε Κάσμαν. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. και ολοκληρώσαμε τις εργασίες μας. Καμιά φορά τελειώνουμε και νωρίτερα. Συμβαίνει και αυτό. Η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 29 Νοεμβρίου, 9 το πρωί με 6.30 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας.